Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή μας συνάντηση είναι αφιερωμένη σε μια δημόσια ακρόαση σχετικά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω θερμά τους τρεις εμπειρογνώμονες που θα συμμετέχουν στη σημερινή συζήτηση και να τους ευχαριστήσω που δέχθηκαν την πρόσκλησή μας. Ο καθηγητής Τζουάχιμ Κούπς, Διευθυντής της Κλόπαν Governance Institute στις Βρυξέλλες, ο οποίος θα επικεντρωθεί στην δεκάχρονη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα διατήρησης της ειρήνης και στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους. Ο πρέσβης κ. Κάρι Κουίνς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρικανική Ένωση και ειδικό απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης, ο δόκτωρ Αλεξάνδερ Μάντελα, βοηθός διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του PUP, ο οποίος θα επικεντρωθεί στο να εξηγήσει την έμμεση προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Προτού τους δώσω τον λόγο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η ακρόαση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για την επερχόμενη έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με το ίδιο θέμα, η οποία θα συνταχθεί στην υποεπιτροπή μας από τον συνάδελφο τον κύριο Βανόρ. Το ισχύο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πρώτη εξέταση της έκθεσης αυτής τον Νοέμβριο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η διατήρηση της ειρήνης είναι μία από τις προτεραιότητες της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας στο πλαίσιο της πολυμερούς στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βασικόν υποστηριχτή τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση στις ειρηνευτικές τους επιχειρήσεις κατά την τελευταία δεκαετία. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμβάλλει μόνο με προσωπικό, αλλά είναι σημαντικός εταίρος της χρηματοδότησης όλων των επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει και δικές της αποστολές υποτυπά για την επιτόπου στήριξη παρόμοιων δράσεων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στο Τσάντ, τον Ταρφούρ και το Κονκόν. Όσον αφορά την Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός προμηθευτής υλικοτεχνικής οικονομικής καθώς και στρατιωτικής υποστήριξης για τις επιχειρήσεις όπως την περίπτωση της Άμυσο, στη Σομαλία και πιο πρόσφατα της αποστολής Φίσμα στο Μάλι. Επομένως, η υποεπιτροπή μας ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον των δύο αυτών σημαντικών σχέσεων και για μια εξέταση των επιτεγμάτων, των αποτυχιών και των μέχρι στιγμής διδαγμάτων από αυτή την συνεργασία. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για τους τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και των κενών στα μέσα και τις δυνατότητες που απαιτούνται για τις αποστολές αυτές. Στόχος μας είναι η εξέβρεση τρόπων για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την διατήρηση της ειρήνης και για την βελτίωση της υποστήριξής μας προς τους άλλους δύο οργανισμούς. Το λόγο τον έχει ο συνάδελφος Βανόρτε. Uh, um, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί σήμερα το απόγευμα μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τη γνώμη επ' αυτού από τους εμπειρογνώμονες και να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, να ακούσουμε κάποιες ιδέες. Βεβαίως και αφετηρία μου είναι το ότι δεν νομίζω ότι είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να κάνει τη στρατιωτική δύναμη, αλλά ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει, να βοηθήσει όσον αφορά την ε, πολιτικού χαρακτήρα παρέμβασή Οπότε είναι ενδεχομένω ε, ε, χρήσιμο κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν χρειάζονται καινούργιε δομέ, δεν απαιτεί ιδιαίτερα χρήματα, δεν επικαλύπτουν δραστηριότητε άλλων θεσμικών οργάνων. Επομένω, το πιο πονηρό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το πιο ευφιέστερο πάντων να, να, να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Και θυμάμαι μια έκθεση που έχω συντάξει στο Κοινοβούλιο αφορούσε κάποια δράση, κάποια πρωτοβουλία για τις νάρκες. Ήταν ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό σαν πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτάξτε τι λέει το, το πόστρο αυτή αφίσα εγώ δεν θα διάλεγα βέβαια αυτή τη φωτογραφία. Title of the report as well, because... Οπότε, κοιτάξτε, ποιος είναι και ο τίτλος, ε, ποιο είναι το θέμα, ε, διότι η διατήρηση της ειρήνης ε, δεν είναι αρκετά ευρύ ως όρος. Καλύτερα να πούμε επιχείρηση υποστήριξης της ειρήνης. Οπότε τελικά το θέμα είναι το τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να ε, βρίσκουμε νέους ρόλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι το θέλουν αυτό, αλλά για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να επισημάνουμε κάποια προστιθέμενη αξία. Πρόεδρε, αυτά προς το παρόν βάζω τελεία και περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις ε, παρεμβάσεις των ε, ειδικών. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βανόρτε και το λόγο έχει ο καθηγητής Τζουάχιμ Κούψ. Ο καθηγητής Κούψ, κύριε Πρόεδρε, εισηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πρώτα πρώτα που με καλέσατε να σας μιλήσω για αυτό το θέμα το οποίο είναι επίκαιρο. Είναι μεγάλη μου τιμή να έρχομαι εδώ. Είναι το θέμα σημαντικό. Με τον συνάδελφο Αλεξάνδρου και τον κύριο Πρέσβη Έχουμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μια ώρα, για να δούμε πρώτα-πρώτα το ευρύτερο τοπίο, να δούμε ακριβώς τι έχουμε πετύχει όσον αφορά την εταιρική σχέση, τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την διατήρηση της ειρήνης. Έχουν γίνει διάφορα, έχουμε ε, την, ε, τη δημιουργία της ειρήνευσης, έχουμε ε, διάφορους, διάφορους τρόπους βοήθειας της υπόθεσης ειρήνη και είναι βασική πολιτική αυτή της διεθνούς κοινότητας του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να σας πω ποια είναι τα τέσσερα σημεία που θέλω να καλύψω σε αυτή την σύντομη μου ε, παρέμβαση. Βεβαίως και μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Πρώτα-πρώτα έχουμε ποιες, είναι οι βασικές προκλήσεις. Ε, έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί την τελευταία δεκαετία. Ε, έχουμε τη θεσμοποίηση, έχουμε την παρέμβαση της κοινότητα, εχουμε έχουμε ε, πάρα πολλά κράτη-μέλη, τα οποία επίσης έχουν προσπαθήσει να βοηθήσουν περισσότερο μετά το 2014. Γιατί μετά το 2014, διότι ελπίζουν ότι μετά από το ότι έχει αποσυρθεί το ΝΑΤΟ από πολλά μέτωπα, υπάρχουν τώρα περισσότεροι πόροι που θα μπορούσαν να ε, παρασχεθούν εις την υποδιατήρηση της ειρήνης. Και θεωρήσαμε ότι έτσι ε, βεβαίως θα υπάρχει συγκράτηση των δαπανών του ΝΑΤΟ. Να δούμε τώρα που δεν τα πήγαμε καλά, ε, πώς μπορούμε τις ελλείψεις που υπάρχουν να τις άρουμε και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μέση διάταξη που θα πρέπει να προσπαθούμε να τηρήσουμε και πώς θα μπορούμε να γνωρίζουμε όλες μας τις δυνατότητες, πώς και το Κοινοβούλιο μπορεί να δραματίσει τον ρόλο που πρέπει και, το, και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Επόμενη διαφάνεια. Να σας τονίσω τώρα ότι ή τώρα ή ποτέ. Αν θεωρείτε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει περισσότερο στη διατήρηση της ειρήνης. Έχουμε σημειώσει σημαντικές πρόοδους όσον αφορά τα επιχειρησιακά. Όπως είπατε και ο Πρόεδρος, είχαμε συνεργασία το 2003 στο Κονγκό, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, το 2006 ε, είχαμε την ΔΑΣΕ, και το 2008 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εκεί που είχατε μία αποστολή παράλληλη με τον ΟΗΕ. Είναι αυτές οι τρεις μεγάλες επιχειρησιακές συνεργασίες. Οπότε βεβαίω είχαν υπάρξει κάποια προβλήματα, αλλά ήταν γενικά χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και βοήθησε τον ΟΗΕ. και σε θεσμικό επίπεδο είχαμε επιτυχίε, πάρα πολύ χρήσιμο γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα εάν αυτό δεν μεταφράζεται σε κάποιο αντίτυπο σε επίπεδο επιχειρησιακό. Οι συναντήσει, ε, ε, τα κοινά θεσμικά δεν πρόκειται να προωθήσουν καθόλου ε, την υπόθεση τη ειρήνης. Αυτά όλα είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Τα τελευταία δέκα χρόνια, από θεσμικών ε, στο θεσμικό επίπεδο δηλαδή, κάναμε πολλά, ξεπνούμε πολλή ενέργεια. Ε, θα πρέπει να δούμε τα πολιτικά ζητήματα και τα ζητήματα των πόρων. Επίση, θα πρέπει να δούμε το ότι υπάρχει εδώ ένα κίνδυνο κόπωσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΟΗΕ. Έχουμε την, ε, μια δεκαετία από τότε που είχαμε την Ιταλική Προεδρία, ένα σωρό προεδρίες και είχαμε την υποστήριξη του σχεδίου τη της ε, ΔΑΣΕ και αυτά όσον αφορά λοιπόν την κοινωνισμό με τις ανάγκες της ΚΕΠΑ, Στα αγγλικά επίσης έχουμε το θέμα της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ. Ε, ξεκίνησε αυτή η υπόθεση τη δεκαετία του 1990. Εκεί από πλευράς ε, ε, ελέγχου και αρχηγίας ε, κατεύθυνση των επιχειρήσεων είχαμε διάφορα προβλήματα ίσως γιατί ε, θα χρειαζόταν περισσότερος διάλογος θα χρειαζόταν περισσότερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ένωσης και ΟΗΕ Ακόμα υπάρχει αντίληψη ότι ακόμα ισχύουν αυτά που ισχύουν το 1993 κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι αληθές Τέλος, θα πρέπει να σας πούμε ότι τώρα έχουμε ένα άνοιγμα, έχουμε μια ευκαιρία. Έχουμε αυτή την εμπροστοφυλακή των 6-7 κρατών μελών, οι οποίοι θέλουν να βρεθούν κάποιοι ρευστικοί τρόποι για να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια καλύτερη ε, προσπάθεια όσον αφορά την διατήρηση της ειρήνης. Βέβαια, πολλές χώρες έχουν μια τέτοια παράδοση ε, είχαμε λοιπόν τη δεκαετία του 1990, αυξήθηκε το βάρος του ΝΑΤΟ, ήταν μια μικρή διακοπή, αλλά παραδοσιακά ευρωπαϊκές χώρες, ε, περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ε, είναι αφοσιωμένες ε, εκτός από το, και εκτός από το ΝΑΤΟ και στη διατήρηση της ειρήνης. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε επομένω την απόσταση των Ευρωπαίων και της Δύσης από τα μέσα τη δεκαετίας του 1990 μετά από την Ρουάντα, τη Σερμπρένιτσα, τη Σομαλία και δεν τα πήγαμε καλά, είχαμε θέματα μένουν αρχηγίας, είχαμε πολιτικά προβλήματα τα οποία ακόμα σοβούν και επίσης είχαμε και κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Κάποιες είναι πιο πολύ φιλικέ στα ΟΝΟΙΕ, κάποιες λιγότερο. Αυτό όμως είναι φυσικό και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε σύγκληση, να έχουμε μια ενιαία φωνή, αλλά βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν και στου κόλπους του ΟΗΕ. Και από τα μέσα μου στα τέλη του 1990, τα κράτη-μέλη εστίασαν την προσοχή τους στο πολιτικό κεφάλαιο και στους πόρους και για τον ΝΑΤΟ και για την ε, αναδυόμενη επιτροπή, ε, ε πολιτική ασφάλεια, εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι το δίλημα τώρα αυτής ε, ΚΕΠΑ, ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια ισχυρή βούληση για αυτόνομη δράση και ξεχωριστό ρόλο της Ένωσης. Αυτό είναι το καλό, κακό, τέλος πάντων είναι άλλη υπόθεση. Αλλά η λειτουργία είναι σημαντική γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ο καλός Σαμαρίτης. Πρόκειται για μια σειρά πολιτικών που έχουμε ασκήσει στο παρελθόν και που βγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι το θέμα της πολυμέρειας ε, από την εποχή του Σολάνα υπήρχε ένας προβληματισμός ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίζει και γι' αυτό και θα πρέπει να συμπλέει με διεθνείς φορείς όπως και με τον ΟΗΕ. Και έτσι ε, και αυτοί οι οργανισμοί γίνονται πιο αποτελεσματικοί. Οπότε αυτής εξ αρχής και ΚΕΠΑ δεν ήταν κάτι τυχαίο, δεν ήταν κάτι αλβριστικό, αλλά ήταν ηθελημένο να προωθηθεί. Ε, είχε να κάνει με τον ρόλο του ΟΗΕ. Θέλουμε επομένως να στήσουμε τον ΟΗΕ, αλλά την άλλη θέλουμε να έχουμε μια ξεχωριστή εικόνα, να ε, προβαλόμαστε σαν ε, αυτόνομη ύπαρξη Βέβαια εδώ πρέπει να προσέξουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και αυτό μας θυμίζει τι έγινε στο, στο Τσάδο το 8 και το ε, 2006 στο, στο Τσάδο. Οπότε, για παράδειγμα, οι πόροι οι οποίοι επενδύονται στην ΚΕΠΑ ταυτόχρονα αφαιρούνται, και στερούνται οι δυνάμεις που και οι πολιτικές που ήδη έτρεχαν, ήδη είχαν ξεκινήσει και θυμάμαι ότι είχα αναμειχθεί με αυτά και θυμάμαι ότι όσον αφορά τις ομάδες μάχης του ΟΗΕ είχε εκεί έπρεπε να αποφασιστεί αν τα, τα, τα στατεύματα εκεί πέρα θα υποστηριζόντουσαν από πόρους της, ε, που θα πήγαιναν κατευθείαν στον ΟΗΕ ή θα τα χρησιμοποιούσαν οι χώρες μέλη. Φαντάζομαι ο Αλεξάνδρ θα σας τα πει καλύτερα. Οπότε νομίζω μην σας για αυτό το σημείο. Και υπάρχει ένα ε, σημείο που πετύχαμε και πρέπει να το υποτιμούμε, δεν ήταν θέμα γραφειοκρατικό, είναι το πώς σιγά σιγά δημιουργήσαμε μια, ένα, μια θεσμικού χαρακτήρα σχέση του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, πέραν του θεσμικού, θα πρέπει και επιχειρησιακά να δούμε πώς θα αποδίδει καλύτερη συνεργασία. Χρειάζεται ε, ισχυρή δέσμευση, χρειάζονται τακτές συναντήσεις, οι διευθύνουσες επιτροπές, όσον αφορά την ασφάλεια, αυτές που συνεδριάζουν ε, κάθε έξι μήνες, μια στις Βρυξέλλες και μια στη Νέα Υόρκη. Και για πρώτη φορά, από το 2012, είχαμε ε, ένα γραφείο ε, αξιωματικού συνδέσμου που συνέβε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ. Και έτσι έγινε διαπραγμάτευση που κράτησε 2,5 χρόνια για ένα σχέδιο δράση, το οποίο τελικά εγκρίθηκε σε ρυθμικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο έγινε και από πλευρά ΟΗΕ. Αυτέ είναι λοιπόν οι θεσμικέ επιτυχίε, αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμούνται. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατικό. Δεν είναι ακόμα ένα έγγραφο. Είναι το τέλος μιας μακράς διαδικασίας που ξεκίνησε τέλος δεκαετίας του 90 και προχώρησε. Και πρόκειται για την πιο στενή θεσμική σχέση όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια. Από πλευράς παραεπιχειρησιακής, και εκεί έχουμε κάποιες επιτυχίες, αλλά και κάποια συμπεράσματα, μαθήματα να αντιλήσουμε και λόγω να είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε την ε, βαθιά σταθερή δέσμευση της Ένωσης όσον αφορά το Σέρμπριτ του ΟΗΕ. Αυτή την ε, ταξιαρχία ταχείας παρέμβασης. Ήταν πολύ υπέρ οι σκανδιναβικές χώρες, είχαμε τις ομάδες μάχες και κάποιοι είχαν πει ότι γι' αυτό το λόγο ε, αφαιρούνται ε, από τις ταξιαρχίες αυτές ε, χρήματα και πάνε στον ΟΗΕ ή το ανάποδο. Και γι' αυτό είπαμε θα πρέπει να δούμε τι συμβατότητες ή ασυμβατότητες υπάρχουν. Ήδη σας είπα τις δύο περιπτώσεις της συνεργασίας, αντλήσαμε από εκεί συμπεράσματα και για τα δύο θεσμικά όργανα, την άριστη πρακτική και έχουμε ευρύ ανταλλαγή απόψεων κατάρτιση, κοινή, κοινό προγραμματισμό σε υψηλό επίπεδο. Από το 2009 βεβαίως, να μην ξεχνούμε, κάτι που δεν είναι μία σύμπτωση. Το 2009 είναι το ορόσημο, τότε που η ΚΕΠΑ ε, από υψίστη προτεραιότητα έγινε λίγο χαμηλότερη προτεραιότητα. Τότε, το 2009, η ΚΕΠΑ ε, από εκεί που ήταν βασικό θέμα γίνεται ένα θέμα πιο light, λιγότερο σημαντικό και το ίδιο φορά και τις σχέσεις επομένω με τον που του οποίου ΔΙΣΚΕΠΑ. Δημιουργία δυνατοτήτων, ε, δεσμεύσεις, Κάποια αυτά που ίσχυαν το, ε, πριν το 9 τώρα δεν υπάρχουν και πρέπει να το θυμηθούμε αυτό αν θέλουμε να ανανεώσουμε την υποστήριξή μας στη μεγάλη αυτονομία. Έχουμε βέβαια πολλά συμπράσματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινεί για το τι πάει καλά και δεν πάει καλά η συνεργασία των δύο οργανισμών. Πάμε τώρα στι αποτυχίε. Ίσως αυτό είναι πολύ απεσιόδοξο σαν έκφραση, αλλά να πούμε τα πράγματα το όνομά του. Έχουμε κάποιε αποτυχίε και πρώτα-πρώτα είναι αυτό ο θεσμικός χαρακτήρας που, έχει, που είναι, ε, είναι κάτι που έχει φτάσει σε βάθος, αλλά δεν έχει φτάσει σε βάθος η, επιχειρησιακή πλευρά της υπόθεσης. Ε, έχουν δεσμευτεί, έχουν αποσυρθεί στην υπόθεση πολλοί αξιωματούχοι, αλλά τελευταία τριετία, τετραετία αυτό δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη υποστήριξη επιτόπου στο πεδίο της δράσης. Τι είναι το σχέδιο δράσης, ε, άλλο το να τα λένε οι γραφειοκράτες και άλλο το να υλοποιούνται όλα αυτά τα προγράμματα σε επίπεδο των μελών, εκεί που υπάρχουν και οι πόροι. Μιλάω για το σχέδιο δράσης, το πιο πρόσφατο που αποφασίστηκε το 2012. Η αλήθεια είναι ότι η υποστήριξη προς τον ΟΗΕ είναι πάρα πολύ επιλεκτική, ανάλογα με το πού προβαλόμαστε περισσότερο, πού θεωρούμε ότι... πού προτιμούμε τέλο πάντων. Γιατί έχουμε και κάποιες εντάσεις όσον αφορά στον διεθνή μας ρόλο σε σχέση με τον ΑΕΑ. Ε, αυτή είναι κάπως ε, εγγενείς αυτές οι εντάσεις όσον αφορά τις φιλοδοξίες και την υποστήριξη. Ας πούμε σε σχέση με την ε, Αφρικανική Ένωση και την Σέρμπρικ, την δύναμη ταχείας παρέμβασης. Μην ξεχνούμε, όταν μιλούμε για συνεργασία, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα επιτυχίας. Όμως, η, αυτή η δύναμη ταχείας παρέμβασης δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε. Ε, ο Καναδά, κάτω χώρες, μετά τη Ρουάντα, μετά τη Ρεμπέντσα, μετά τη Σομαλία και, και από άλλες χώρες, όχι μόνο από Καναδά. Και κάτω χώρες για να αποτρέψει ε, άλλες γενοκτονίες θα αφορούσε τον Αγία και μόνο για ταχεία παρέμβαση σε περιπτώσεις ε, γενοκτονίας. Και σας πενθυμίζω ότι στον χάρτη του ΟΗΕ, στο άρθρο 43 και 45, προβλέπονται η στρατηγική δράση του ΟΗΕ και αυτή η ταξιαρχία είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει για να δημιουργήσουμε κάποιο είδους στρατός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δράση της ταξιαρχίας στην Αφρική έξι φορές. Ε, βοηθήσαμε τη δημιουργία δυνατοτήτων, καινούργιων δυνατοτήτων για την ε, Αφρική, γιατί και εκεί δημιούργησαν μετά κάποιες ε, ε, δυνάμεις οι Αφρικανοί, θα σας τα πει και ο κύριος Πρέσβες. Οπότε ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία της ταξιαρχίας για να έχουμε αυτήν την την δύναμη ε, τη στρατιωτική από πλευρά Αφρικανών. Και πολλές φορές οι οργανισμοί είναι μακρόβιοι. Σε αυτή την περίπτωση όμως εξέπνευσε κατά κάποιο τρόπο, ήρθε στο τέλος της ζωής του κύκλου ζωής της αυτή η δύναμη και οπότε χρειάστηκε να έχουμε τριπλή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ. Αυτοί οι τρεις φορείς ασχολήθηκαν και εκεί κατέληξε. Αλλά πέραν αυτού δεν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αρνητικοί, γιατί ακόμα ε, έχουμε πάρα πολλά να διδαχτούμε από την εμπειρία εκείνη όσον αφορά τη δημιουργία δυνατοτήτων, την Αφρικανική Ένωση σε σχέση με τον ΟΗΕ, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τριμερείς ε, επαφές ε, ακριβώς για την δημιουργία παραδικών δυνατοτήτων αλλά βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν οι πόροι και πολλές φορές η... εάν κάποιος ασχολείται στον ένα οργανισμό αυτό σημαίνει ότι υπονομεύει τον άλλο. Άρα είναι θέμα πολιτικής προτίμησης το ποιον οργανισμό κανείς θα στηρίξει. Τέλος, έχουμε κάποια παγιά προβλήματα τα οποία ε, αφορούν την, της, της ειρήνης, έχουμε ακόμα πολύ σκεπτικισμό όσον αφορά το σύστημα αρχηγίας και ε, το επιτελικό τέλο πάντων όσον αφορά την ηγεσία των έλεγχων πλευρά ΟΗΕ. Ακόμα υπάρχουν πολλά θέματα επιμέρους να ρυθμιστούν. Ακόμα δεν έχουν επιληθεί όλα, αλλά υπάρχει πρόοδος. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν προσπάθειες για τη ειρήνης. Στην ναι, όχι πάντως υπάρχει μια μονάδα ευρωπαϊκή. Εκεί είμαστε πρότυπο. Αλλά οι, οι άλλοι στον ΟΗΕ, εκτός αυτής της υπηρεσίας, θεωρούν ότι είμαστε ενόχληση γιατί θα έπρεπε κανείς να ενεργεί είτε από τη μία πλευρά του ελληνικού και από την άλλη και ότι θεωρούν παράξενο το ότι υπάρχει τέτοια υπηρεσία ευρωπαϊκή μέσα στο ΝΑΤΟ. Έχουμε τα θέματα τώρα πολιτική εντολή και πολιτική βούληση. Ε, αυτό είναι ένα προβληματισμός στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει η εντολή να μελεταθεί καλύτερα, θα πρέπει το Συμβούλιο ασφαλεία, να εμπλέκεται περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία αλλά αυτό θα πρέπει να το επιλύσει ο ΟΗΕ. Πάντως όταν λέμε ΟΗΕ έχουμε δύο μόνιμα μέλη που λένε α, η... έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αλλά βέβαια τον μπαλάκι είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων και αυτοί θα πρέπει να ξεδιαλύνουν την κατάσταση. Έχουμε εδώ και ανταγωνισμούς μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ, αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι γίνεται με τους οργανισμούς αυτό γίνεται και στην Αφρικανική Ένωση και αλλού. Υπάρχουν επίσης τέτοιοι ανταγωνισμοί και σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, όμως δεν είναι αγεφύρωτο το χάσμα. Επίσης, τον ανταγωνισμό που ανέφερε ο εισηγητής, πάντοτε είναι ένα καυτό θέμα τα χρήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύει ούτως ώστε να μπορέσει να τηρήσει τα όσα έχει υποσχεθεί σχετικά με την ΚΕΠΑ. Ας πούμε, αυτό ισχύει και όσον αφορά την ε, την, την πολιτική άμυνα κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν είναι αστήρευτη η να καλύψουμε όλους τους οργανισμούς, όλες τις δράσεις. Επίσης υπάρχει ισχυρή προτίμηση οι Ευρωπαίοι να προτιμούν το ΝΑΤΟ γιατί εκεί ασκούν περισσότερη επιρροή. Περισσότερη επιρροή στο ΝΑΤΟ παρά στον ΟΗΕ εκτός από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά σκεφτείτε ποιοι στέλνουν στα ειρήνη. Στο Μπαγκλαντέ, στην η Ινδία, το Πακιστάν, όχι οι Ευρωπαίοι. Εκείνοι στέλνουν στα άρα εκείνοι επηρεάζουν το σύστημα στο, περιθώ... στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Άρα, επομένω, προτιμούν οι οργανισμοί που έχουν δυτικό στυλ από του Ευρωπαίου. Τέλο, τι θα γίνει μετά το 2014. Αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία, ούτω ώστε να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα όσα ισχύαν προηγουμένω για την για την διατήρηση ειρήνης από πλευρά ΟΗΕ. Έχουμε την Χάισαφ ε, που είναι η πιο βασική δέσμευση της Ένωσης προς τον ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Στρατή ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες αποστολές. Πάντως, η ΚΕΠΑ τώρα είναι πιο εξελιγμένη. Έχει επένδυση περισσότερα μέτωπα παρά στην εποχή του Σολάνα. Επομένως, αυτό σημαίνει θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των στρατευμάτων, ανάπτυξη, εμπειρία και άρα κάποιες χώρες ίσως θελήσουν να ασχοληθούν περισσότερο με την υπόθεση αυτή. Γιατί υπάρχουν και κάποιες μικρότερες χώρες, ιδίως Σκανδιναβοί, που στα σοβαρά τώρα σκέφτονται πώς μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο. Αυτό με σε επίπεδο επιμελητία, σε επίπεδο προσφορά ελικοπτέρων και άλλους τρόπους να σε να βοηθήσουν. Άλλα ζητήματα τώρα τα οποία πρέπει να επιληφθούν οι δυνατότητες που θα πρέπει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλει να αναβαθμιστεί ο ρόλο της. Θυμηθείτε τι έγινε στο μαλλι. Για να αποδειδούν περισσότερο χρειάζεται πιο έντονος διάλογος και υπάρχει το συνεχές θέμα που εκρεμεί για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. και πολλά διακυβεύονται από πλευρά πολιτική σε σχέση με το σχέδιο δράση από πλευρά των μελών. Το κοινοβούλιο τι μπορεί να κάνει. Ε, στο χέρι του το τι θα κάνει για τι δυνάμει διατήρηση τη ειρήνη. Χρειάζεται πιο έντονο διάλογο από πλευρά κοινοβουλίου με την DPKO και επίση την Υπηρεσία Ασφάλεια και Ειρήνη του ΟΗΕ. Εδώ, στι Βρυξέλλε. μπορεί να αναπτυχθεί διάλογο. Περισσότερο εδώ παρά στον, στη Νέα Υόρκη. Και επίσης θα πρέπει να διευκολυνθεί με τον κύκλο των φύλων ο διάλογο που ονομάζεται η επιστροφή τη Ευρώπη στην διατηρήση τη ειρήνη. Θα πρέπει να συνεχιστεί ε, το να προβάλλεται, το να ακούει τη δυνατή φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την ΚΕΠΑ και να έχει κάποια αυτονομία και να είναι και αυτή υπαρκή αυτή η πολιτική. Εδώ θα βάλω τέλεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή και τον λόγο να έχει ο πρέσβης κύριος Κάρις Κουίνς. Uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα προσπαθήσω να συμπληρώσω την εισήγηση του Γιώργεν, ιδιαίτερα για την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας δύο λόγια για την εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Ιδιαίτερα στο τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι Ό,τι κάνουμε σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση εμπίπτει στην κοινή μας ε, εταιρική σχέση, την κοινή ε, στρατηγική ε, Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε στην διάσκεψη κορυφής που έγινε το 2007 στη Λισαβόνα και θέσπισε αυτή τη στρατηγική. Επανεπικυρώθηκε το 2010 στην Τρίπολη και θα είναι και αντικείμενο τη επόμενη διάσκεψης κορυφής που προβλέπεται να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς, ε, όπου ήδη ξεκινάμε την εργασία μας με, το, με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και τα μέλη της Αφρικανικής Ένωσης για το μέλλον της εταιρικής σχέσης. Είναι εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο υπήρους, αλλά εργαζόμαστε με υπάρχοντα ε, δημοσιονομικά μέσα. Το βασικό είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά για τη Βόρεια Αφρική υπάρχει και η εταιρική σχέση γειτονίας και από του χρόνου θα υπάρχει και άλλο ένα μέσο, το Παναφρικανικό πρόγραμμα που για πρώτη φορά θα δώσει ένα γεωγραφικό μέσο που καλύπτει ολόκληρη την Αφρική και βέβαια υπάρχουν και άλλα μέσα που αναγράφονται εκεί, δηλαδή οι διμερείς συμβολές, συνεισφορές των κρατών μελών μας προς την Αφρική. Η ίδια στρατηγική αποτελείται από οκτώ θεματικές εταιρικέ σχέσεις. Κάθε μία εξ αυτών έχει τους δικούς της στόχους και πρόγραμμα δράσης. Και θα εστιάσω στην υπαριθμόν 1 που είναι η εταιρική σχέση ειρήνη και ασφάλεια. Θέλω να τονίσω αυτές οι μεμονωμένες εταιρικές σχέσεις συνδέονται μεταξύ τους και όλος ιδιαίτερος οι δύο πρώτες που βλέπετε εκεί, δηλαδή ειρήνη και ασφάλεια και δημοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα συνδέονται αναπόσπαστα και η προσέγγιση της Ένωσης προς την ε, διάσκεψη κορυφής του Απριλίου, εμείς προτείνουμε στους Αφρικανούς συναδέλφους αυτές οι δύο εταιρικές σχέσεις να συνδυαστούν σε, ένα, σε μια εταιρική σχέση που θα ε, τετλοφορείται ειρήνη και δημοκρατία και θα αναγνωρίζει ότι βασικό πρόβλημα, ε, βασική, η ρίζα μάλλον πολλών προβλημάτων στην Αφρική είναι το θέμα της διακυβέρνησης. Η εταιρική σχέση ειρήνης και ασφάλειας, θα έλεγα, ε, έχει τρεις βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι να βελτιωθεί ή να αυξηθεί ο διάλογος ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε κοινέ θέσεις και να εφαρμόσουμε κοινέ προσεγγίσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Αφρική, αλλά να καλύψουμε και την Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια θέματα, όπως η τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, ε, ξέπλυμα χρήματος και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι να στηρίξουμε την Αφρική στην, ε, στην δημιουργία και την, ε, της, αρχιτεκτονικής, της αφρικανικής αρχιτεκτονικής για την ειρήνη και την ασφάλεια και το τρίτο είναι να δούμε ποια είναι η πιθανή χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που, ε, των οποίων ηγείται η Αφρική. Το βασικό μέσο που χρησιμοποιούμε είναι η Αφρικανική Διευκόλυνση για την Ειρήνη και δημιουργήθηκε το 2004. Αυτά που κάνουμε με το Ταμείο Ανάπτυξης και τη Διευκόλυνση για την Ειρήνη στην Αφρική είναι διαφορετικά. Δεν εμπίπτουν όλα όμως μέσα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτά τα μέσα. Τι είναι λοιπόν η αρχιτεκτονική, ε, αφρικανική μάλλον ε, αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας. Όταν ε, δημιουργήθηκε η Αφρικανική Ένωση το 2002, άλλαξε μια βασική της προσέγγιση που ήταν η αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών της με την αρχή της μη αδιαφορίας για τα εσωτερικά και εισήγει την αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας από αυτές τις βάσεις. Δημιούργησε το, Συμβούλιο Ασφαλείας και Ειρήνης της Αφρικανικής Ένωσης ως το βασικό όργανο, το οποίο βοηθείται από μια στρατιωτική επιτροπή. Επίσης υπάρχει μια ομάδα των σοφών που αποτελείται από διακεκριμένες αφρικανικές προσωπικότητες και είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην διαμεσολάβηση καθώς και ένα ε, ε, παναφρικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που δίνει πληροφορίες για πιθανές περιοχές σύγκρουσης. Όλα αυτά υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα. Στη συνέχεια προβλέπεται η, η δύναμη μια αφρικανική ένοπλη δύναμη stand-by. Στόχος είναι να είναι επιχειρησιακή το 2015 θα υπάρχουν ε, πέντε περιφερειακές ταξιαρχίες που θα αποτελείται κάθε μία από 5.000 ε, στρατό με δυνατότητες ε, ταχείας ανάπτυξης. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν δηλαδή σύντομα σε περιπτώσεις κρίσης. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα, η ειρήνη δυστυχώς κοστίζει. Εδώ βλέπετε τα ποσά. Το ένατο και δέκατο ταμείο για την ειρήνη έχουν δώσει περίπου 1.200, ε, εκατομμύρια ευρώ ε, τα τελευταία 7 χρόνια. Από το 2007 έχουμε έναν ε, μηχανισμό έγκαιρης ανταπόκρισης, ένα μικρό ποσό, ώστε να βοηθήσουμε την Αφρικανική Ένωση να αντιδράσει γρήγορα σε τομείς όπως είναι η πρόληψη των συγκριούσεων ή η μεσολάβηση. Και χρηματοδοτούμε με αυτά τα 17 εκατομμύρια διάφορες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αφρική. Έπειτα, η δημιουργία της αφρικανικής αρχιτεκτονικής ειρήνης και ασφάλειας, για τη δημιουργία δηλαδή θεσμικών δυνατοτήτων για την ειρήνη και την ασφάλεια, στήριξη της κατάρτισης και μέσω αυτής και τη δημιουργία της αφρικανικής ένοπλης ε, δύναμης. Και ο πιο σημαντικός, το πιο σημαντικό τμήμα είναι ένα δις, έχει πάει στην οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων στήριξης της ειρήνης. Εδώ μια διαφάνεια που δείχνει τις βασικές επιχειρήσεις σε στήριξη της ειρήνης στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Οι δύο βασικές για την Αφρικανική Ένωση είναι η Άμισομ στη Σομαλία με 17.700 στρατιώτες και η Αφίσμα στην Κεντρική ε, Αφρικανική Δημοκρατία όπου προτείνεται να περάσουμε από τους 750 στρατιώτες σε 3.500 ε, τους επόμενους μήνες, αλλά ακόμα μελετάται αυτή η πρόταση. Έπειτα έχουμε 8 επιχειρήσεις του ΟΗΕ για την στήριξη της ειρήνης, 84.000 κόσμος, προϋπολογισμός 5,5 δις δολάρια. Ο προπολογισμό για την Αμισόμ και για, την, ε, για τη Σομαλία δηλαδή και την ε, Κεντρική ε, Αφρική είναι περίπου ένα δις. Δηλαδή σύνολο όλων των επιχειρηματικών επιχειρήσεων είναι 6,5 δις δολάρια ετησίως. Τεράστιο ποσό. Ας το συγκρίνουμε με τον προπολογισμό της Αφρικανικής Ένωσης. Ο ετήσιος προπολογισμός τους, ο διοικητικός, είναι κάτω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα κόστος τελείως δυσανάλογο σε σχέση με τις ε, δυνατότητες της Αφρικανικής Ένωσης. Δεν μπορεί να το καλύψει. What can we pay from the African Peace Facility? Τι μπορούμε να πληρώσουμε εμείς από τη διευκόλυνση. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό ή πυρομαχικά, αλλά μπορούμε να πληρώσουμε το κόστος ανάπτυξης, ε, πιστούς, ε, ιατρικά κτλ. Ετήσιοι μισθοί στο κάθε στρατό δίνονται, μηνιαίοι μάλλον μισθοί, δίνονται από τις ε, συμβαλόμενες χώρες. Ο ΙΕ παρεμβαίνει, συμβάλλει με την διοικητική μέρημνα και διάφοροι άλλοι δωρητές διμερείς, κυρίως οι ΙΠΑ που έχουν διμερείς, διμερείς συμφωνίες με διάφορες χώρες. Προσπάθησα να συνδέσω την ε, Αφρικανική Ένωση με τον και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα, η σχέση της ε, Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση είναι μέσω της εταιρική σχέσης ειρήνης και ασφάλειας. Και μια παρόμοια εταιρική σχέση υπάρχει, έχει συναυθεί ανάμεσα στον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση. Και ανάμεσα σε όλους υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς οι, οι αποστολές στήριξης της ΚΕΠΑ μπορούν να στηρίξουν τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ. Και υπάρχει ένα σχετικό σχέδιο που έχει συναυθεί το 2011. Τώρα, επιτόπου Πρέπει να πω ότι ε, το τρίγωνο αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε έμπιστοι εταίροι τόσο της Αφρικανικής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη ε, αναθεώρηση της ΑΜΙΣΟΜ, ε, της επιχείρησης της Σομαλία. Και ο στρατιωτικός σύμβουλος της δικής μου αντιπροσωπείας εκλήθη να συμμετέχει και συνδέθηκε πλήρως, ε, συμμετείχε πλήρως στις συζητήσεις για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η αποστολή Άμισομ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα καλείται να είναι μέρος ε, του σχεδιασμού από, το, από τα πρώτα στάδια, από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού κάθε επιχείρησης. Φυσικά πρέπει να τονίσω ότι δεν λειτουργούμε εν κενό. Ε, όλα αυτά είναι τμήμα της γενικής μας προσέγγισης. Έχουμε μια γενική προσέγγιση για το κέρας της Αφρικής, για το Σαχέλ, για το Ανατολικό Κονγκό και την Κεντρική Αφρική. Να σας δώσω το παράδειγμα της Σομαλίας, όπου εργαζόμαστε σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας, σε επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας, σε επίπεδο ασφάλειας βέβαια, η Αμισόμα όπως σας ανέφερα υπάρχει και η αποστολή κατάρτισης που εκπαιδεύει τους Σομαλούς για τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας. Υπάρχει η UCAP Nestor για τις ε, θαλάσσιες ικανότητες και η UNAFOR που καταπολεμεί την πειρατεία στις ακτές ε, της ανοιχτά της Σομαλίας. Και όλα αυτά εντάσσονται σε μια συνολική προσέγγιση. Πρόσφατα, όπως μάλλον θα γνωρίζετε, υπήρξε και η διάσκεψη New Deal για μια νέα συμφωνία για τη Σομαλία που προσπάθησε να διερευνήσει το μέλλον το, από την αναπτυξιακή πλευρά, από την άποψη της οικοδόμησης κράτους στην χώρα αυτή και δεσμεύτηκε για 8 δις 8 δις δεσμεύτηκαν από τους διάφορους δωρητές για το μέλλον, για την ανάπτυξη του, ενός μέλλοντος για τη Σομαλία. Θα έλεγαμε λοιπόν ότι στην Αφρική πλέον ε, η Αφρικανική Ένωση είναι αξιόπιστος και σημαντικός εταίρος. Όταν μιλάμε μια φωνή, ο υπόλοιπος κόσμος ακολουθεί. Μπορείτε να δείτε την περίπτωση της Σομαλίας, του Σουδάν, όπου η Αφρικανική Ένωση βασικά θέσπισε την ημερήσια διάταξη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ακολούθησε αυτήν την ατζέντα. Τώρα, το Συμβούλιο Ασφάλειας και Ειρηνή της Αφρικανικής Ένωσης είναι ε, ένα όργανο με μέγα κύρος. Για παράδειγμα, αν γίνει πραξικόπημα σε οποιαδήποτε χώρα στην Αφρική, να δώσω το παράδειγμα του Μαλή πέρυσι, μέσα σε 24 ώρες συνεδρίασε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας, καταδίκασε το πραξικόπημα και εντός 48 ώρων ξανασυνεδρίασε και ε, ε, έθεσε σε αναστολή το Μαλί από την ε, Αφρικανική Ένωση. Το ίδιο έγινε και με τη Γουινέα Μπισάου. Έχει βάρος, έχει κύρος δηλαδή σε ολόκληρη την Ήπειρο. Και όπως σας έλεγα, ε, η Είναι αλήθεια ότι οι συγκρούσεις στην Αφρική διαρκώς μειούνται τα τελευταία χρόνια. Είναι επίσης γεγονός ότι το τελευταίο χρόνο υπήρξε μια ιδιαίτερη αναταραχή στο Σαχέλ, η συνέχεια του προβλήματος στη Σομαλία και οι, οι, εξεγέρσεις στην κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία αλλά και στο Ανατολικό Κονγκό και χρειάστηκαν πολλοί πόροι για να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα όλες αυτές οι κρίσεις και είναι νομίζω αξιέπαινη η Αφρικανική Ένωση που κατάφερε να το κάνει αυτό και να διατηρήσει ηγετικό ρόλο. Όπως σας είπα δεν μπορεί να το κάνει μόνη της και η Αφρικανική Διευκόλυνση για την Ειρήνη αναγνωρίζεται ως ένας από τους βασικούς ε, υποστηριχτές φορείς και αναγνωρίζει φυσικά και τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι τώρα οι προκλήσεις. Η στήριξή μας προς την Άμισον φέτος φτάνει περίπου τα 205 εκατομμύρια ευρώ και ίσως ε, αληθεύει αν πούμε όταν το δούμε ως ένα πρόγραμμα βοήθειας γιατί χρησιμοποιούμε βοήθεια, κονδύλια βοήθειας, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα βοήθειας που έχουμε οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι ε, τεράστιο βάρος για μας και παρά τις προσπάθειές μας, πέρα από μας, τον ΟΙΕ, τους, τις υπάρχουν ελάχιστοι άλλοι διεθνείς εταίροι που συμμετέχουν στη στήριξη της Αφρικανικής Ένωσης. Δεύτερον, πρέπει περαιτέρω να τελειοποιήσουμε και να καθορίσουμε το καταμερισμό εργασίας των διαφόρων φορέων. Ο ΙΕ και η Αφρικανική Ένωση πρέπει να βελτιώσουν τα πράγματα όταν δηλαδή θα ε, σκεφτήκαμε την διευκόλυνση, ε, δεν προβλέψαμε ότι θα στήριζε μια επιχείρηση όπως η Άμισομ ή μάλλον ότι η Αφρικανική Ένωση θα έπρεπε να συντηρήσει μια επιχείρηση της κλίμακας της Άμισομ για έξι χρόνια και πάνω με την πιθανότητα να χρειαστεί να συνεχίσουν για τουλάχιστον ακόμα τρία χρόνια. Προβλεπόταν ανέκαθεν σίγουρα από εμά ότι η Αφρικανική Ένωση και οι αφρικανικές επιχειρήσεις οι ειρηνευτικές θα ήταν συντομότερες και ότι θα υπήρχε μια μετάβαση προς ε, τον ΟΗΕ. Αλλά με την άμεσο δεν έγινε αυτό. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της σχέσης ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση και τις περιφερειακές οργανώσεις που θα πρέπει να ενισχυθεί και να ε, τελειοποιηθεί. Έπειτα, πλήρης επιχειρησιακός χαρακτήρας της ε, αφρικανικής αρχιτεκτονικής ε, ειρήνης και ασφάλειας και η δημιουργία ένοπλων αφρικανικών δυνάμεων. Βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται στην κεντρική δημοκρατία, αφρικανική δημοκρατία. Τα πράγματα χειροτερεύουν κάθε μέρα και αργούν πάρα πολύ, αργούν πάρα πολύ να ε, κινητοποιήσουν την αφρικανική ε, δύναμη που χρειάζεται εκεί. Από τη δική μας πλευρά χρειάζονται πολλαπλές παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τα κράτη-μέλη και καλύτερο συντονισμό, Αλλά ακόμα και αν γίνει τέλειο συντονισμό, είναι γεγονό ότι οι προπολογισμοί μα, τα κονδύλια και οι διαδικασίε βρίσκονται σε διαφορετικά κανάλια και υπάρχουν κενά. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε τα λεφτά τη Άμισομ να τα πάρουμε και να πάμε στο UCAP Nestory ή από την αποστολή κατάρτιση και να τη βάλουμε αλλού. Δεν πάει έτσι και γι' αυτό και δημιουργούνται κενά σε αυτά που κάνουμε και σίγουρα χρειάζεται να ενισχύσουμε περαιτέρω το συντονισμό μας εδώ και επιτόπου. Κοιτώντα λοιπόν προς το μέλλον θα έλεγα ότι οι τρεις βασικοί τομείς που βλέπετε εδώ είναι οι ίδιοι βασικά όπου δουλεύουμε δηλαδή και τώρα σε όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να τονίσω τα πρώτα σημεία, ότι χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο για την μοιρασιά του οικονομικού βάρους τόσο από αφρικανικές χώρες, διότι θα πρέπει να βρουν, να, να μπορέσουν και εκείνες να συγχρηματοδοτήσουν αυτές τις τεράστιες επιχειρήσεις, αλλά και από τον ΟΙΕ και άλλους νέους, αλλά και παραδοσιακούς δωρητές. Και έπειτα Πρέπει να δουλέψουμε για στρατηγικές εξόδου, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πού πάμε και πού πάει και η Αφρική. Αυτή είναι η τομή που ε, εργαζόμαστε. Υπάρχει όμως ένα άμεσο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και οι συνάδελφοί μου εργάζονται από αυτού. Είναι το 10ο ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που εκπνέει στο τέλος αυτού του έτους, ενώ το 11ο δεν θα αρχίσει να ισχύει παρά μόνο το 2015. Το 2014 μένει στο κενό δηλαδή. Πρέπει να δουλέψουμε τώρα σε αυτό και όπως είδατε και στο Ναϊρόμπι πριν από λίγες μέρες, ο πόλεμος κατά της Αλσεμπάμπ δεν είναι ένας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Αμισόμ πρέπει να συνεχιστεί ε, το 2014 και πιο πέρα και πολύ πιθανότατα θα πρέπει και να ενταθεί. Ε, αλλά αυτό δημιουργεί τεράστιο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αποστολής. Αυτό το, αυτή η διαφάνεια είναι το website μας, είναι ένα κοινό website που έχουμε με την Αφρικανική Ένωση. Βάζουμε όλη μας τη δουλειά εδώ, σε, αυτή, τη, σε αυτό το site. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρέσβη και το λόγο να έχει ο κύριος Αλεξάνδρ Μάτελα. Dear Mr. Chairman. κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση να σας μιλήσω εδώ σήμερα. Επέλεξα να εστιάσω στο ακαδημαϊκό κάπως θέμα της ε, έμεσης ε, προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ειρήνης. Θα το κοιτάξω από ακαδημαϊκής ε, γωνίας. Έχω τρία βασικά τμήματα στην παρουσίασή μου. Καταρχάς, να εξηγήσω το τι σημαίνω. Τι σημαίνει ακριβώς αυτή η έμεση προσέγγιση. Τι εννοώ με αυτό. Να προσπαθήσω να εξηγήσω την τάση την οποία θεωρώ ότι διαφαίνεται. Και τρίτον, εξηγήσεις για να δούμε κατά πόσον στέκουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα και τέλος θα θέσω το ερώτημα του κατά πόσον όντως υπάρχει λογική, υπάρχει σκοπός. Και θα χρησιμοποιήσω το έργο που έκανα μαζί με τον συνάδελφό μου, ε, τον κύριο Μαρέινεν, ο οποίος κάθεται στην απέναντι άκρη της αίθουσας, μέρος ενός βιβλίου για την διατηρήση της ειρήνης στην Αφρική. Θα ξεκινήσω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, τι σημαίνει έμεση προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κρίση της ειρήνης. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα συμπλήρωνε το έργο άλλων διεθνών οργανισμών, είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη, το Βορειοδυτικό Σύμφωνο, την Αφρικανική Ένωση. Η συνεργασία λοιπόν αυτή δεν είναι κάτι το καινούριο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι η ακριβής κατανομή των εργασιών αλλάζει. Και αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την διαχειρισιακή στάση της, ε, την επιχειρησιακή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται λοιπόν με τις επιχειρήσεις ε, υπό την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν στα αριστερά μία εικόνα όπου προβάλλεται το σήμα της ε, EU4. Θα μπορούσα να έχω επιλέξει και άλλη επιχείρηση. Ή θα μπορούσα να έχω επιλέξει και την επιχείρηση του, των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Λίβανο, όπου βασικά Ευρωπαίοι στρατιώτες συμμετείχαν. Αυτό που έχουν από κοινού λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις, οι πιο παλιές ε, της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, είναι ότι είχαν μια στεναρή πολιτική βούληση πίσω από την εντολή. Η χρήση δηλαδή βίας θα πρέπει να περιοριστεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τις ε, αεροπορικές επιδρομές, όπως για παράδειγμα στο Τσάντ, και στις αποστολές αυτές ήταν πραγματικά εξαιρετική η ικανότητα η επιχειρησιακή από πλευρά ε, των ευρωπαϊκών ε, στρατευμάτων και από πλευρά τακτική και από πλευρά τεχνολογία και τεχνολογική εξειδίκευση. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριαρχούσαν ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σκέλος και έτσι σημαντικά έπαιζαν ένα αποτρεπτικό παράγοντα το οποίο είχε φυσικά άμεσα μια συνέπεια σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Οι νέες τώρα επιχειρήσεις και πα, που έχουν ξεκινήσει πιο πρόσφατα, βλέπετε στο δεξί τμήμα της διαφάνειας μια εικόνα όπου ευρωπαϊκές δυνάμεις εκπαιδεύουν τις ε, δυνάμεις στο Μαλί και στη Σομαλία η σχετική επιχείρηση σε ό,τι αφορά τα σύνορα στη Σοσαχέλ, στο κέρας της Αφρικής. Σε όλα λοιπόν αυτά τα νέα περιβάλλοντα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ουσιαστικά αναπτύσσουν το δυναμικό. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν εκπαιδευτικούς σκοπούς αντί να δημιουργούν άμεσα μέσω του αποτρεπτικού τους χαρακτήρα ένα σύστημα ασφάλειας βοηθούν πλέον έμεσα υποβοηθώντας τη γενικότερη ασφάλεια. Αυτή είναι λοιπόν η τάση των τελευταίων ετών. Για όσους ε, από εσά ε, έχουν κάνει στρατηγικές σπουδές, θα καταλαβαίνετε φυσικά ότι αυτό το, το όρο τον δανείζαμε από τον Sir Base Little Heart, ε, Βρετανό ιστορικό. Όπου αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι η στρατηγική πάντα έχει ως στόχο της την μεταφορά, την ξερίζωση κάποιων τέτοιων στοιχείων. Άρα η διατήρηση της ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ως σκοπό να παραμείνουν πολλά στρατεύματα επιτόπου, αλλά να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου την ειρήνη θα την διατηρούν άλλοι. Να υποδείξω επίσης, μετά από αυτά που ακούσαμε και προηγουμένως από τους συναδέλφους, ότι αυτή η τάση προς μια έμεση προσέγγιση συμπληρώνεται από τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο διευκόλυνσης ε, για την Αφρική αναφέρθηκε να προσθέσω ότι ο Αλεξάνδρ Ρόντος, ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Αλσαμπάμ. Αυτό τι σημαίνει ότι αν διευρύνουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα θα δούμε ότι αυτή η έμεση προσέγγιση ξεπερνά τα όρια της διατήρησης της ειρήνης όπως να ορίζεται. Γιατί αν κάποια κράτη μέλη αποφάσιζαν για παράδειγμα να υποστηρίξουν τους αντάρτες στη Συρία και αυτό θα αποτελούσε ε, ένδειξη της ισχύω αυτής. Αλλά είμαι ακαδημαϊκός και θα σας εξηγήσω αναγκαστικά γιατί παρουσιάζεται αυτή η τάση. Έξι αίτια ουσιαστικά εγώ εντοπίζω. Κάποια εξ αυτών είναι αλληλοσυνδεόμενα και σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Να υποδείξω καταρχάς ότι αυτό έχει νόημα σε ό,τι αφορά την τοπική ιδιοκτησία. Αφρικανική λύση για αφρικανικά προβλήματα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο επιχείρημα ότι πρόκειται για αποδοτική χρήση των χρημάτων. Γιατί τα νέα αυτά προγράμματα, τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι πιο φθηνά, σημαντικά πιο φθηνά σε σχέση με τις παλιές επιχειρήσεις. Μιλάμε για προϋπολογισμό 10 έως 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για παράδειγμα η επιχείρηση στο Τσάντ που δεν ήταν καν μεγάλη ήταν κινούνταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη Λιβύη, για παράδειγμα, ρωτιόμαστε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται μόνο στην ε, αρρωγή για την, τους συνοριακούς ελέγχους. Γιατί, αν θέλουμε να κρατήσουμε την ειρήνη στη Λιβύη, χρειαζόμαστε 30 έως 120.000 ε, στρατεύματα ανάλογα με την υπολογισμό. Και προφανώς κανείς δεν θέλει να δώσει τόσο στρατεύματα επιτόπου εκεί. Τρίτο αίτιο σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Συζητώντας τις παλιές επιχειρήσεις, δίνω έμφαση σε αυτό το χαρακτήρα τον αποτρεπτικό. Αυτός είναι ο πυλώνας της στρατηγικής και της λογικής των επιχειρήσεων. Αλλά αυτός ο αποτρεπτικός χαρακτήρας έχει νόημα μόνο ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η στρατιωτική απειλή. Δεν μπορεί να παραμείνει αυτό για πάντα. Αντιθέτω αυτέ οι επιχειρήσει αναπτύξή δυναμικού με πιο ελαφρύ αλλά πιο ε, μακροπρόθεσμο αποτύπωμα, αν θέλετε, είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν η φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε και να αναρτούμε την Ευρωπαϊκή Θερμαία, ο πιο φθηνός τρόπος είναι αυτός. Τέταρτο αίτιο, που το βλέπουμε και στη σχετική βιβλιογραφία. Σε κάποιο βαθμό είναι μεγαλύτερη η ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την οικονομική, τα οικονομικά συμφέροντα των οικονομικών δυνάμεων στο κέρας της Αφρικής και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και αυτό ασφαλώς έχει να κάνει με την στρατηγική τους διάσταση και έτσι μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι θα μπορούσε κανείς να αναθέσει στα τοπικά, στους τοπικούς φορείς τέτοια καθήκοντα προκειμένου να ανακύψουν πλατφόρμες που θα υποστηρίξουν ε, τις ευρωπαϊκές πολιτικές τα επόμενα χρόνια. Πέμπτο αίτιο, το οποίο θα ήθελα να σας επισημάνω, κάτι που το έγραψε και το έχει εξηγήσει ο συνάδελφός μου Λύση Σιμών, επί Μακρόν. Η ανάπτυξη δυναμικού φαίνεται ότι είναι το μοναδικό έργο επί το οποίο μπορούν να συμφωνήσουν πλέον οι Ευρωπαίοι, γιατί μπορούμε φυσικά να πούμε από την επιχείρηση Σερβάλ, για παράδειγμα, θεωρήσαμε ότι ήταν καλή την επιχείρηση από το Παρίσι, ενώ η κρίση στο Σαχέλ αναπτυσσόταν επί σειρά ετών, αργά. Τελικό αίτιο. Το τέλος της ε, διαχείρισης της κρίσης. Και στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια θα σας εξηγήσουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν εδώ στο γράφημα το σύνολο των συνεισφορών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυμερείς τέτοιες επιχειρήσεις ειρήνευσης και σταθεροποίησης. Είτε μιλάμε για δράση του ΙΕ και το καθεξής. Εξαιρούνται οι εθνικές οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις συνασπιμού. Μιλάμε δηλαδή για συνεισφορές καθαρά σε πολυμερή τέτοια θέματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ποιες ήταν οι τάσεις ε, στα τέλη του ψυχρού πολέμου. Μεγάλη αύξηση κατά τον πόλεμο στη Ιγκοσλαβία, στο, στην κρίση του κοσυχοπεδίου και μια δεύτερη μ, κορύφωση όταν ε, το η επιχείρηση στο Αφγανιστάν και μετά μια πτωτική τάση από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς ασφαλώς, αλλά και με το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Γιατί αυτή η αύξηση σε ό,τι αφορά το τη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων έχει να κάνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σχετική περίοδο και την παράδοση. Αν λοιπόν σιγά σιγά ξεθυμένει αυτό το παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει και η σχετική πολιτική για την ασφάλεια και την ειρήνευση. Σας υποσχέθηκα ότι θα κλείσω με μία ερώτηση. Έχει νόημα αυτή η τάση. Ναι, έχω να σας πω, αλλά έχω να βάλω και κάποια κάποια, κάποιες υποσημειώσεις. Η ανάπτυξη λοιπόν δυναμικού για να διατηρείται η ειρήνη από άλλους έχει νόημα και από πλευράς οικονομικής και πολιτικής γιατί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ειρηνευτικές διαδικασίες χωρίς όμως να εκτίθεται υπερβολικά. Αυτό είναι ιδανικό για περίοδους ε, λιτότητας. Αλλά τρία στοιχεία να αναφέρω Καταρχάς, ε, συχνά δίνεται αυτό το ζήτημα ανάπτυξης δυναμικού σε ομοιοπαθητικές δόσεις. Είναι σαφές ότι πολύ συχνά υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούμε σε ψευδείς πόθους. Μπορεί να μπορούμε να αναρτήσουμε την Ευρωπαϊκή Σημαία σε μια περιοχή σύγκρουσης στέλνοντας 50 συμβούλους, αλλά δεν είναι πολύ πιθανό ότι αυτό πραγματικά θα περιορίσει την κρίση στην χώρα εκείνη. Δεύτερο, δεύτερη σημείωση. Αν δημιουργηθούν πιο ικανές ε, τοπικά δυνάμεις ασφάλειας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πιο αποτελεσματικέ τέτοιε αστυνομικέ και στρατιωτικές δυνάμει είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί δεν ακολουθούν πάντα δημοκρατικά, δημοκρατικές ε, πολιτικές. Άρα έχουμε την επιρροή που θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε απαραίτητα όλα και ασφαλώ αυτά μπορεί να μα γυρίσουν μπούμεραν. Τα τεράστια ποσά σκεφτείτε που έχουν ε, δώσει οι Αμερικανοί για το στρατό της ε, Αιγύπτου. Αλλά αναρωτιέμαι τι ακριβώς επιρροή αγοράζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι σαφές αυτό. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι μόνο πρόβλημα της Αμερικής, να κοιτάξετε το website της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας, να επιλέξετε το χάρτη των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και μετά να επιλέξετε το εικονίδιο για την ε, επιχείρηση στη Γουινέα Μπισάου. Θα δείτε ότι η διεύθυνση δεν ισχύει πλέον δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ αν αυτό είναι σύμπτωση. Τελευταίο στοιχείο. Υπάρχει επίσης ένας κίνδυνος να παρανοήσουμε και να θεωρήσουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις ανάπτυξης δυναμικού είναι οι πραγματικές επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, όντως είναι μια σωστή και εύλογη λύση. Αλλά σε κάποια άλλες περιπτώσεις η προστασία των ευρωπαϊκών αξιών μπορεί να απαιτεί πραγματικές δυνάμεις, πραγματικά στρατεύματα. Άρα θα πρέπει να γίνεται μια επιλογή και να υπάρχει αυτή η επιλογή και να ξέρουμε ότι δεν εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη δυναμικού επειδή είναι το μοναδικό πράγμα αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το λέω κλείνοντας να σας επιστήσω την προσοχή στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι τα στρατεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες περιπτώσεις ε, αποδεκατίζονται. Δηλαδή μειώνοντας τον αριθμό τους και αυτό μειώνει ασφαλώς και την ικανότητά τους. Αλλά να πρωτοπροσέξουμε αυτό για να μην μείνουμε χωρίς όπλα στα χέρια μας εάν τα πράγματα πραγματικά ξεφύγουν. Τον κύριο δεν ξέρω αν ο συνάδελφος ο κύριος Βανόρτεν έχει κάτι να απαντήσει ή να σχολιάσει. No, I, I found it all... Uh, Πάρα πολύ συναρπαστικά είναι αυτά που ακούσαμε και από τους τρεις ε, εισηγητές. Πάντως το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι πάρα πολύ απίλαψα αυτά που ο κύριος Μάτελα πάντως παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι έχουμε αυτό το την μεταβολή, την μείωση της βούλησης, της διάθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να εμπλακεί. Και αυτό δεν το φαντάζονταν κανείς αν άκουγε μόνο τις συζητήσεις εδώ στο Κοινοβουλίο ή σε άλλα θεσμικά όργανα ευρωπαϊκά. Δηλαδή το πώς έχει η σε αλλα θεσμικα ευρωπαικα δηλαδη το πως εχει η οποία δεν συμβαδίζει ε, με την ρητορική και οι στρατιωτικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα λόγια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και για αυτό και ε, θέλανε και αυτή τη συνάντηση του Δεκεμβρίου για το Συμβούλιο Ασφάλειας, όμως, ε, Συμβούλιο Άμυνα, συγγνώμη, αλλά στην πραγματικότητα άλλο συμβούλιο όπως γνωρίζετε, ε, δεν ξέρω αν γίνονται επίτηδες όλα αυτά ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία είπατε ε, μας προβλημάτισαν πάρα πολύ. Ε, όλους εμάς οι οποίοι ε, είμαστε αναφαντών υπέρ του να έχει σε αυτά τα θέματα μεγαλύτερη πιο σημαντικό την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τις ε, εξελίξεις για την έμεση προσέγγιση νομίζω ότι κάποια πράγματα τα παραλείψατε δηλαδή πρώτα πρώτα την αλλεργία την αλλεργία ως προς τα να έχουμε κάποιες απώλειες από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γιατί Ξέρουμε ότι ε, η ο κόσμος τώρα, γίνει είναι αλλεργική σε αυτές τις ε, απώλειες και άρα θα ήθελαν και την πίτα ο Λάκερ και το σκύρο χορτάτο να αφορά τις δραστηριότητες του, τις στρατιωτικές. Τώρα γιατί έχει εμπλακεί στις ε, επιχειρήσεις διαχείρισης των συνόρων, στη Λιβύη, ε, και το, το, το, το μίσο έκανε. Μα ναι, μα δεν, δεν, δεν, το θέλανε. Και οπότε γι' αυτό και απελπισμένα προσπαθούμε να βρούμε κάποιο δικό ρόλο, αλλά ήταν και ανεπιθύμητοι και δεν θέλαμε κι εμεί τόσο πολύ. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να ρωτήσω και του τρει είναι το εξή. Με όλα αυτά τα δεδομένα, τι θεωρείτε ότι είναι το πιο χρήσιμο που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας κατά μέρος τα λόγια τη φιλοδοξία του ρόλου του ως παγκοσμίου παράγοντα των ε, στρατών της Ένωσης πέρα από όλα αυτά, αν θα ήθελε να κάνει κάτι χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς ε, υποστήριξη της ειρήνης ε, στον ΟΗΕ, στην Αφρικανική Ένωση, τι είναι το πιο χρήσιμο. Μόνο να δίνει λεφτά. Ευχαριστώ τον κύριο Βανόρτεν. Κύριος Φίσας, απορτέραν Θέλει να πάρει τον λόγο. Ο κύριος Κάλερ. Thank you for the very... Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κυρία Γκόμες, για τα όσα ενδιαφέροντα μας παρουσιάσατε. Το 2004 ήρθα στο Κοινοβούλιο. Και από τότε η διαδρομή ήταν πάρα πολύ μακρά και όλα αυτά τα οποία επιτύχαμε από τον Αύγουστο του 2004 και μετά είχαμε 150 τότε ε, ε, πρόσωπα στο, στο, στον σε εμβριακή κατάσταση να δουν τι θα γίνει στην ευριακή κατάσταση τέλο πάντων αποστολή εκεί, για να μπορέσουν να υποστήξουν ε, τι προσπάθειε εκεί. Αλλά από τότε πέρασαν πάρα πολύ, γιατί κοιτάξτε τώρα έχουμε 17.000 στην Σομαλία. Άρα, τι να αποδείξουν έχουμε για το ότι έκανε τη διαφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εταιρική τη σχέση, τη συνεργασία τέλο πάντων με την Αφρικανική Ένωση. Πάντω παραμένουν οι προκλήσει, παραμένουν τα νέα προβλήματα και χρειάζεται μια προσέγγιση συνεπή. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Φτύνουμε τον κόρφο μας. Όλοι. Για το ότι δεν έχουμε εμπλακεί στην εκπαίδευση αυτών που αντιμετωπίζουν τους τρομοκράτες στον Αερόμπι. Τέτοια επομένω προσέγγιση χρειάζεται. Όπω είπαν και οι μιλητέ για την ε, Γίνα της το τη αποστολή τη ΚΕΠΑ, την αποσύραμε ενώ θα έπρεπε μάλλον να έχει ενισχυθεί, θα έπρεπε να έχει ε, πάρει καινούργια κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε το πραξικόπημα, αλλά μετά μετά στράφηκε στους υπεύθυνους για λόγους εσωτερικών ε, αντιπαλωτήτων Νιγηρίας, Αγγόλας. Κύριε Πρέσβη, θα ρωτήσω για την ε, Γουίνια Μπισάου. Εκεί που βλέπουμε να έχουμε όλα αυτά τα δίκτυα τρομοκρατών, τα δίκτυα των εγκληματιών που εμπλέκονται με τους δε, ε, ε τι γίνεται στον Παναμά, στον κόλπο της Γουινέας, την πειρατεία. Τι χρειάζεται που να κάνουμε για να πετύχουμε ασφάλεια στη θάλασσα και συγκεκριμένα εκεί στον κόλπο της Γουινέας. Και αυτό δεν καίει μόνο τους Αφρικανούς αλλά και εμάς. Για τη Λιβύη τώρα. Τζέφρι, Τζέφρι, ξέρεις τι πιστεύω για αυτό που είπες, αλλά εσείς κύριοι συμφωνείτε. ότι θέλετε ή δεν θέλετε να υπάρχει αποστολή της ΚΕΠΑ στη Λιβύη. Γιατί τώρα σιγά σιγά ξεκίνησε δραστηριότητα τέτοια διαχείριση των συνόρων, ενώ γνωρίζουμε ότι ε, αυτά που κάνουμε είναι ανεπαρκή και ήρθαν πάρα πολύ αργά γιατί τελικά ε, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ε, εκπαιδευμένος στρατός. Ενώ δεν υπάρχει. Κάτι παραστηριοτική είναι μόνο εκεί. Τα κράτη-μέλη όμως αυτό πρέπει να κάνουν. Όμως τα κράτη-μέλη αυτό το οποίο θέλουν είναι τα πράγματα να συνεχιστούν όπως είχαν και πριν. Business as usual. Να πουλάνε στον Καντάφη, να, αντί για τον Καντάφη να πουλάνε αυτά που πουλούσαν εις την νέα κυβέρνηση. Τι τους νοιάζει περιφερειακή ασφάλεια. Να τώρα όπλα από τη Λιβύη πάνε στη Συρία. Οπότε η Λιβύη εστράφει στο ΝΑΤΟ. Και στο ΝΑΤΟ βέβαια θα εκπροσωπούνται οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες που θα κληθούν τώρα να αναλάβουν δράση. Αλλά δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί προφανώς οι χώρες οι οποίες ε, υπό την αιγύδα του ΝΑΤΟ θα εμπλακούν, πρόκειται να πληρώσουν. ΝΑΤΟ και όχι και πάει. Επομένως, κύριε Κουίντς, πέστε τι πιστεύετε τι γίνεται με την Αφρικανική Ένωση, μια που έχουμε αυτή τη, το επίσημο αίτημα της Λιβικής κυβέρνηση, μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό. Τέλος δε, για το Μάλι. Για το Μάλι. Να, μια περίπτωση ότι για οικονομικού λόγους τα κράτη-μέλη δεν παρενέβησαν, δεν ενεπλάκησαν. Για πετε μας εσεί πώ το βλέπετε. Είναι θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να επιληθεί στο επόμενο Συμβούλιο. Τα έχουμε πει σε πολλές εκθέσεις. Και έχουμε και την πιο πρόσφατη έκθεση για ΝΑΚΟ. Επίσης, κανόνα της εμπλοκής. Όλο και περισσότερη υπεργολαβία ούτως υπήν έχουμε τώρα. <coughs> Όχι μόνο για την Αφρική. Αλλά έχουμε ιδιωτικές εταιρείες. Μισθοφόρων. Τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ε, κατηγορίες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για χρήση όπλων κλπ. Ο Σφίσα, από την ΤΕΡΕ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο εισηγητής για την έκθεση της Επιτροπής Συνεργασίας. Ήταν πάρα πολύ εξαιρετικά τόσο επανόλυωση έλαβαν τον λόγο. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μάτελερ βασικά, αλλά μπορεί να απαντήσει οποιοδήποτε άλλο θέλει από τους εισηγητές. Είπατε ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει κυρίως η Ευρώπη είναι να εκπαιδεύσει αφρικανικές δυνάμεις. Πότε θέλετε έχουμε ένα πραγματικό αφρικανικό στρατό ο οποίο θα μπορεί να αναλάβει το έργο της πρόληψης συγκρούσεων στην Αφρική Άλλο δηλαδή κάποιος να εκπαιδεύεται, να εκπαιδεύει, να ενημερώνει, γιατί φοβάμαι ότι αυτός ο Αφρικανικός στρατός έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του ή και αν ποτέ σχηματιστεί. Ευρωπαϊκέ δυνάμει, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, θα πρέπει έτσι και αλλιώ να είναι εκεί επί τόπου. Α, κοιτάξτε, στο Μάλι. Είχαμε ΟΗΕ, είχαμε Γάλλους, οι Γάλλους υπό την αιγίδα του ΟΗΕ θα μπορέσουν κάποτε να ε, πάρουν τις τύχες στα χέρια τους οι Αφρικανοί. Yeah. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη δέσμευσή μας με την Αφρικανική Ένωση θα σας το πω και ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Αποστολής για το Παραφρικανικό Κοινοβούλιο. Οι Αφρικάνοι εταίροι μας μας λένε τακτικά ότι σε αυτές τις οκτώ εταιρικέ σχέσεις στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική, ο τομέας και της ασφάλειας και της άμυνας λειτουργεί καλύτερα από όλους. Και αυτό δεν ε, μας προκαλεί έκπληξη γιατί πάντα υπάρχει μια συγκεκριμένη κρίση και δημιουργούνται συγκεκριμένες ανάγκες. Και τότε μπορούμε να αποφασίσουμε με ποια μορφή μπορούμε να βοηθήσουμε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις αυτές. Καταρχάς, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της Αφρικανικής Ένωσης ε, δραστηριοποιούμαστε και αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι κάτι πολιτικό εκφυταίο αφενός. Κατά δεύτερον, επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να βγούμε από το σύστημα, από ένα μηχανισμό του συστήματος, από το σύστημα των μηχανισμών ad hoc και να βρεθούμε σε μια κατάσταση που διαρκώς θα βοηθούμε την Αφρικανική Ένωση και θα αναπτυχθεί μία δύναμη η οποία θα είναι stand-by, θα είναι έτοιμη να παρέμβει για να εφαρμόσουν τις δικές τους λύσεις, αφρικανικές λύσεις για αφρικανικά προβλήματα. Ναι, ωραία. Στρατιώτες, ε, δομές, ε, εξοπλισμός, όλα αυτά χρησιμοποιούνται και δίδονται για να, μπορεί να μπορούν να δράσουν αυτό είναι και πολιτικά αποδεκτό στην Ευρώπη. Να πούμε ότι με αυτή την μόνιμη διάθεση και προθυμία να σας συνδράμουμε με εμπειρογνωμοσύνη, με υποδομές και το να μεταβούμε εμείς με τα δικά μας στρατεύματα θα πρέπει να είναι κάτι όχι μόνο επικουρικό αλλά και κατά περίσταση, μόνο όταν είναι αναγκαίο. όταν είναι αναγκαίο και για τα δικά μας συμφέροντα και όταν μας ζητείτε ρητά. Θα προτιμούσα όμως με εκπαίδευση και υποδομές να βοηθήσουμε προκειμένου επί της αρχής στην Αφρική να μπορούν να λαμβάνονται αφρικανικά μέτρα. Να επανέλθω όμως στην κρίση στη Λιβύη. Αφενός ε, δραστηριοποιηθήκαμε και δώσαμε μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια. Βοηθήσαμε τους πρόσφυγες ε, στα σύνορα της Λιβύης, στην ε, Αίγυπτο, στην Τινησία. Και δώσαμε φάρμακα, δώσαμε εφόδια στην πολιορκημένη αυτή πόλη. Αλλά είχαμε προγραμματίσει να υπάρχει μια δύναμη stand-by, η οποία θα είχε ως σκοπό να προστατεύσει με στρατιωτικό τρόπο την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Δηλαδή δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφαλίζουμε με στρατιωτική δύναμη. Αυτό όμως τελικά μπλέχτηκε στο ΟΗΕ γιατί αντιστάθηκαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Άρα θεωρώ ότι το θέμα δεν ήταν μια κόπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΙΕ θεωρώ ότι ένα πολιτικό, ένας πολιτικός κικαιώνας, όπου τελικά δεν υπήρχε επιθυμία από κάποιος να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με boots on the ground, με συγκεκριμένες δυνάμεις. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι δεν υπήρχε αυτή η επιθυμία να ασφαλιστεί στρατιωτικά αυτή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθεια. Πώς θεωρείτε λοιπόν, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ικανότητες των ε, Ηνωμένων Εθνών στο μέλλον να αναπτύξουν και να αποδεχτούν μια συνολική προσέγγιση προκειμένου για παράδειγμα να δεχτούν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δίδουμε ανθρωπιστική βοήθεια και όταν είναι απαραίτητο μπορούμε με τα δικά μας στρατεύματα στα πλαίσια του ΟΗΕ να προστατεύσουμε τα άτομα αυτά που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. Τι γίνεται λοιπόν με τις σχετικές συζητήσεις, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και το λόγο έχουν τώρα οι εμπειρογνώμονες μας. Θα ξεκινήσω αντίστροφα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Αλεξάνδερ Μάτελαρ. Thank Σας ευχαριστώ που μας κάνετε αυτές τις καλές ερωτήσεις ε, για να απαντήσω στον κύριο Φανόρδεν. Τι είναι το πιο χρήσιμο, το πιο ωφέλιμο που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά, αυτά που έχουν ήδη γίνει είναι λογικά από αρκετές απόψεις. Εγώ σκόπιμα σας παρουσίασα ποιες ήταν οι συνεισφορές για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΗΕ για να σας πω ότι οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να πείξουν τι δυνάμει του σε διάφορα πλαίσια και όλα αυτά τα πλαίσια συνεπάγονται κάποια πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα φάση είναι, όπως είπατε κι εσείς, ότι η θεωρία δεν συνάδει πάντα απαραίτητα με την πράξη. Άρα νομίζω ότι τα βασικά μηνύματα που έχω να σας αποστείλω είναι να εξετάσουμε το τι συμβαίνει πραγματικά σε οργανισμούς άμυνας για να αποφασίσουμε προς τα που οδεύουμε. Το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο ενδεχομένω να είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο. Υπό τον όρο ότι τα κράτη-μέλη δεν θα χρησιμοποιήσουν το θέμα της ε, ενισχυμένης ε, συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συγκαλύψουν ενδεχομένω το τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Κατά πόσον ε, μπορούμε να ελπίζουμε και να καλοδεχτούμε έναν Αφρικανικό στρατό σύντομα. Δεν είμαι μάγος και δεν μπορώ να μοντέψω. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο άμεσα. Να σας επιστήσω την προσοχή όμως στην περίπτωση του Τσάντ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγει την πιο μεγάλη αυτόνομη επιχειρησή της το 2008-2009. Τότε το Τσάντ ήταν στο χείλος της προς τα... της, αν θέλετε, μιας έκρηξης προς τα έσω. Κοιτώντας τι έγινε και στο Μάλι, για παράδειγμα, φέτος, συγκρίσιμη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγε στρατιωτική επιχείρηση, η οποία προβλήθηκε με πολύ αρνητικό τρόπο και είχε αρνητική διαφήμιση για διάφορους λόγους, αλλά βλέπουμε ότι η στρατιωτική στρατηγική στρατηγική εξίσωση έχει πλέον μεταβληθεί δραματικά και το τσάντ ήταν ο πιο βασικός παράγοντας που συνεισέφερε στο να δραστηριοποιηθούν τα γαλλικά στρατεύματα στις αρχές του έτους στο Μάλι. Άρα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν θέλουμε ικανές στρατιωτικές ε, δυνάμεις, αυτές χρειάζονται σε τελική ανάλυση μία ισχυρή οικονομία. Πώς δημιουργούμε λοιπόν Αφρικανικό στρατό, Α, εκπαιδεύοντας τον, ε, τους Αφρικανούς ή δημιουργώντας μία πιο λειτουργική αγροτική πολιτική. Δεν ξέρω απομακρυνόμαστε και θα έπρεπε να απομακρυνθούμε από το μοντέλο της συνεργασίας ad hoc. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αρνητικά. Αλλά το κρίσιμο είναι να ξέρουμε προς τα που πηγαίνουμε. Και στην παρούσα φάση θα πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι στο πιο υψηλό πολιτικό επίπεδο οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοιτούν προς τα έσω προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα της Ευρωζώνης και στην παρούσα φάση υπάρχει πολύ περιορισμένο περιθώριο για να εξεταστεί το τι συμβαίνει γενικότερα στον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ κρίμα, γιατί όπως ξέρουμε ο κόσμος μεταβάλλεται ταχύτατα. είναι πολιτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στα πιο υψηλά επίπεδα. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό με ξεπερνάει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και το λόγο έχει τώρα ο πρέσβης κύριος Κάριν Πένς. Well, let me also address the question of what, what should we be doing. I να προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω στο τι θα πρέπει να κάνουμε. Στην παρουσίαση που έκανα ήθελα να τονίσω ότι η εταιρική σχέση ειρήνης και ασφάλειας είναι μία μεταξύ άλλων και φυσικά θα μπορούσα να μιλήσω και για τις υπόλοιπες, αλλά θέλω να εξορροπήσω αυτή την εικόνα που ίσως έδωσα, την εντύπωση που έδωσα ότι η ειρήνη και η ασφάλεια κυριαρχεί στα όσα κάνουμε με την Αφρική. Δεν ισχύει αυτό. Όταν όμως ε, άρχισε τη θητεία η νέα Επιτροπή τη Αφρικανικής Ένωσης υπό την ε, προεδρία του δόκτωρος Ζούμα της δόκτωρο Ζούμα, είπε εκείνη ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε τα όσα κάνουμε στην ειρήνη και την ασφάλεια που είναι πάρα πολλά με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπα νωρίτερα για την επερχόμενη κοινή διάσκεψη κορυφής εδώ στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την δημοκρατική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να το τοποθετήσουμε δίπλα στα όσα κάνουμε για την ειρήνη και την ασφαλή. Είναι αλήθεια, όπως είπε ο κ. Γκάλερ, ότι από πολλές απόψεις η ειδική σχέση ειρήνης και ασφάλειας λειτουργεί καλύτερα γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις στη διακυβέρνηση και άρα συγκρούσεις. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα βέβαια και αυτό είναι τμήμα της ε, συνεργασίας μας με τη νέα Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης. Κάνουμε περισσότερα για τις εκλογές, προσπαθούμε να προωθήσουμε του διάφορου χάρτε για τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπω γνωρίζει ο κ. Γκάλερ, συνεργαζόμαστε με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, την Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα, όπω είπα, υπάρχει αυτή η σύγκληση διαφόρων κρίσεων. Όταν δηλαδή καίγεται το σπίτι πρέπει να σβήσει πρώτα τη φωτιά για να μπορεί να κάνει τη πιο μακροπρόθεσμη δουλειά. Σίγουρα χρειάζεται να φτιάξουμε περισσότερα. Τώρα, αν θα υπάρξει Αφρικανικό στρατό. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα υπάρξει αυτή η δύναμη stand-by, αφρικανική δύναμη stand-by, από τις πέντε ταξιαρχίες που σας είπα. Η Επιτροπή έκανε μια πρόταση για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και τα σαφή προγράμματα που έχουν εντοπίσει στη Βαλή και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία ανάπτυξης, ανάπτυξης δηλαδή στρατευμάτων να δημιουργήσουν μια ε, δύναμη άμεσης ανταπόκρισης της κρίσης. Θα είναι η αρχή για την ε, δύναμη αυτή τη stand-by, την ετοιμοπόλεμη. Δεν μπορώ τώρα βέβαια και να ε, βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να σας δώσω μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά σίγουρα από τη δική μας πλευρά μέσω των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μέχρι το 2015 όντως να υπάρχουν αυτές οι πέντε ετοιμοπόλεμες ταξιαρχίες. Αλλά βέβαια πρέπει να δουλέψουμε και σε εθνικό επίπεδο και η κυρία Γκόμες ανέφερε τη Γουινέα Μπισάου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, ότι στις συζητήσεις για το τι θα κάνουμε με τη Γουινέα Μπισάου και πρέπει να σας πω ότι είχαμε εξαιρετική κοινή αποστολή Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική Ένωση, ΟΗΕ, κοινότητα πορτογαλόφωνων ε, ε, χωρών και τώρα την Φραγκοφωνία και προσπαθούμε να πιέσουμε τα διάφορα μέρη προς τις εκλογές και επιστροφή στη δημοκρατία. Αλλά φυσικά η Γουινέα Μπισάου κυριαρχείται από την εγκληματικότητα και κυρίως από το εμπόριο ναρκωτικών. Η Αφρική και η ECOWAS μας κατηγορούν εμάς. <laughs> Είναι ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα στροφή. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι είναι που καταναλώνουν τα ναρκωτικά, δεν είναι οι Αφρικανοί πράγμα που δεν αληθεύει και ότι ούτε οι Αφρικανοί είναι αυτοί που χειρίζονται το εμπόριο των ναρκωτικών. Ε, δεν είναι και αυτό τελείως αληθινό. Ε, ε, είναι αλήθεια ότι επηρεάζονται από το εμπόριο ναρκωτικών. Δουλεύουμε για τη θαλάσσια ασφάλεια, για τις διαδρομές, τους δρόμους της κοκαίνης. Πάντως, αν θέλουμε να έχουμε μόνιμη ειρήνη στη χώρα αυτή, θα πρέπει να ε, ξαναφτιάξουμε τους θεσμούς από την αρχή και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της εγκληματικότητας που καταλήγει τα πάντα και τον στρατό. ρόλος του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να πω ότι το ΝΑΤΟ είναι σχετικά περιθωριακό σε σύγκριση με την Ένωση. Εντάξει, υπάρχει το, το, τα υπόλοιπα της Λιβύης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτησε διαφορετική άποψη εκεί. Δεν είχε ενωμένη φωνή, αλλά σίγουρα οι χώρες είχαν διαφορετική άποψη για το στρατηγό Καντάφη και την κατάσταση εκεί. Και αυτή ως απόϊχος συνεχίζεται. Ενδιαφέρονται για να αναπτύξουν τις σχέσεις τους, αλλά η Αφρικανική Ένωση ίδια είναι κάπως ψυχρή. Κρατάει απόσταση. Και έπειτα δεν έχω ιδιαίτερο σχόλιο να κάνω για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και του ρόλου του ΟΗΕ. Η ανθρωπιστική βοήθεια σε περιπτώσεις ε, συγκρούσεων είναι πάντα πολύ δύσκολη. Να σας ε, αναφέρω το Σουδάν ως παράδειγμα. Μιλήσατε για 150 ανθρώπους ε, που συμμετείχαν στην αρχική επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης στον Νταρφούρ. Για μας ήταν κάτι που μάθαμε. Ήταν μάλλον μια μαθητεία, γιατί ό,τι κάνουμε στην Αμισόμου τα μάθαμε από, το δικό μας, από τα δικά μας λάθη στον Ταρφούρ. Σήμερα υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις ειρηνευτικές του ΟΗΕ στο Σουδάν και στο βόρειο, νότιο Σουδάν. 25.000 στρατός Τεράστια προσπάθεια. πρέπει να σας πω ότι η Αφρικανική Ένωση ηγείται της πολιτικής διαδικασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ε, ε, ε, σχετικά επικρατεί ειρήνη σε σχέση με το παρελθόν. Το πετρέλαιο ρέει, οι χώρες συνομιλούν μεταξύ τους και είναι ένα καλό παράδειγμα όπου η Αφρικανική Ένωση επιβεβαίωσε την ηγετικό της ρόλο και ο ΙΕ τη στήριξε όχι απόλυτα, γιατί τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν συμφωνούν στα πάντα για το τι πρέπει να κάνουν στο Σουδάν, αλλά εν πάση περιπτώσει και με τη δική μας στήριξη, γιατί μπορέσαμε να στηρίξουμε το πάνελ ε, υψηλού επίπεδου υπό τον πρόεδρο Μπέκη μέσω της, του μηχανισμού έγκαιρης ανταπόκρισης, σήμανε αυτό τη διαφορά. Και για να επανέλθω στο θέμα Τη δυνατότητας ε, παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας δεν καταφέρνουμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο Νταρφούρ αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε πρόσβαση λόγω της ασταθούς στρατιωτική κατάστασης. Παρότι δηλαδή είναι εκεί 35.000 άνθρωποι στι δύο χώρες, ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να παραδώσουμε ε, την ανθρωπιστική βοήθεια που θα θέλαμε ο καθηγητής, ο κύριος που πρέπει να πω ότι κατέθεσε μια πρόκληση που πρέπει να κερδίσουμε. Η τώρα ή ποτέ από ό,τι έχω αντιληφθεί μας έχει πει. Ο κύριος Κουβς; Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ερώτηση. Πιστεύω σε μια ισχυρή Ευρώπη. Ισχυρή και πά. Και ισχυρό ΟΗΕ. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ΟΗΕ όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης. Άλλωστε, όλα τα κρατημερανία μου και στον ΟΗΕ και στα σχήματα τα περιφερειακά που βεβαίως ε, μπορούν να βοηθήσουν την παγκοσμία ειρήνη. Οπότε αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μια ε, βοήθεια, μια συνεργασία χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους, χωρίς επιφυλάξεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες αποστολές που μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά μόνο η Ευρώπη. Βέβαια, δεν αρκεί η οικονομική προσπάθεια. Και να μην ε, βέβαια ε, υπερτιμούμε τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. 7 δις ξοδεύτηκαν για το Αφγανιστάν σε 4-5 μήνες από τις ΗΠΑ. Ε, Άρα χρειάζεται εμπλοκή και οικονομική αλλά και πρακτική, λειτουργική για την έμεση προσέγγιση. Μα από το 2003-2006 δύο αποστολιστές ΚΕΠΑ βοηθήσαμε στο Κονγκό τον ΟΗΕ, σε αυτό το παράδειγμα, αυτό ίσχυσε η ε, έμεση συνεργασία. Και έχουμε και άλλες δύσκολες αποστολές, πέραν του Κονγκό. Βεβαίως μεγάλη εκεί σύγκρουση, χειρότερη γη έγινε με τον καιρό και ε, κάποιους μήνες βοηθήσαμε εκεί πέρα άμεσα τον ΟΗΕ. Όμως εδώ πέρα έχουμε δύο πτυχές στο πρόβλημα. Αυτοί που έχουν κριτικάρει ε, τον ΟΗΕ ότι είναι αδύναμος. Μα για σκεφτείτε, τους βοηθάει κανένας. Είπα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε αυτή την έμεση βοήθεια με τις αποστολές της ΚΕΠΑ. Βοηθάνε. Όμως έτσι αδυνατίζει ακόμα περισσότερο ΟΗΕ, διότι κατά κάποιο τρόπο ε, πάμε λίγους μήνες εκεί, φεύγουμε, τα προβλήματα ανακύπτουν και πάλι, οπότε αυτό εκθέτει τον ΟΗΕ. Αυτό υποβαθμίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ. Ή θα έπρεπε να έχουμε αφήσει κάποιους ε, και αφού έφυγε μεγάλο όγκο τη αντιπροσωπεία μα εκεί, τη δύναμη μα εκεί, ή να έχουμε βοηθήσει αλλιώ άμεσα τον ΟΗΕ. Για τι προσπάθειε λοιπόν ασφάλεια και ε, ειρήνη. Για τον ISF, λίγο πιο απεσιόδοξα εδώ είναι τα πράγματα. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία το 2003, ε, άρχισε να τρέχει το 2010, γίνανε πολλά, δυνατότητες δημιουργήθηκαν και πάμε τώρα για, για, για, για, πιο, για κομβική μερομηνία του 2015. Άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα τα πάνε. Οι βόρειες ταξιαρχίες, οι νότιες ταξιαρχίες, έχουμε κάποιες εκεί πέρα διαφορές. Θα χρειαστεί χρόνος. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές, πολλοί παράγοντες, πολλοί που ανταγωνίζονται. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που τώρα βοηθούν τη δημιουργία δυνατοτήτων στην ε, Αφρική. Σκεφτείτε τι έχουν κάνει οι ΙΠΑ ε, παράλληλα με τον ΝΑΤΟ, παράλληλα με τον ΟΗΕ, γιατί έχουμε κάποια κρατημέλη τα οποία σε εθνικό επίπεδο δρούν εκεί σε επίπεδο εθνικής ε, δημιουργίας ε, δυνατοτήτων, κάτι το οποίο έχει να κάνει βέβαια με, με, με φιλοδοξίες εθνικές, δεν είναι οι καλοί Σαμαρίτες. Όμως χρειάζεται κάποιο του συνέπεια, συνοχή, κάποιο συντονισμό. Άλλος υπάρχουν προβλήματα. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστεί το ISF σε κάθε περίπτωση ε, ξεχωριστού capacity building, ξεχωριστών παραγόντων, ε, βορείων, νοτίων. Σε κάποιες περιπτώσεις είπαμε ότι μέχρι το 2009 είχαμε το Σέρμπρικ το οποίο βοηθούσε, αλλά θα έπρεπε να συντονιστούν, να συνδυαστούν 16 χώρες. εκεί στην Αφρική και το πρόβλημα δεν ήταν τα χρήματα. Όταν άρχισε η δημιουργία δυνατήτων από τον ΟΗΕ ε, δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα. Έπρεπε να υπάρχει συνεργασία υπηρεσιών ε, και αντί του να δαπανώνται, να αναδιασπαθίζονται χρήματα, έπρεπε να υπάρχει συντονισμός, ε, συνεννόηση διαφορετικών υπηρεσιών. Άρα το θέμα εδώ είναι η διαβίβαση πληροφοριών, η μετάδοση κάποιων γνώσεων, εμπειρίας. Απλώς τώρα προσωπικού για αυτές τις δυνάμεις που εφημερεύουν κατά κάποιο τρόπο, που είναι στο stand-by. Όλα γίνανε εκεί. Υπάρχουν δομικά προβλήματα εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα και είναι ένα εργαλείο βιώσιμο, χρήσιμο. Και έχοντας αυτή τη ε, δύναμη που εφημερεύει, δεν είναι αυτό καμιά πανάκια γιατί ο ΙΕ είναι ο μόνος αμερόληπτος οργανισμός που μπορεί να αναπτύσσεται σε συγκρούσεις εκεί που οι τοπικοί έχουν ο καθένας τα δικά τους συμφέροντα. Και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τις δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης όπως ήταν στο Μαλία. Και εκεί οι τοπικοί οι ηγεμόνες έχουν τα δικά τους συμφέροντα αυτοί που παρεμβαίνουν εκεί. Ε, αυτό μπορεί να τυφασευθεί μόνο με τον ΟΗΕ. Για τη Λιβύη τώρα, κύριε Γκάλα, το ζήτημα εκείνο της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και της στρατιωτικής υποστήριξης, όπως εγώ κατάλαβα, όπως έμαθα, είναι το ότι το θέμα ήταν το τι θα κάνει η εκεί υπηρεσία του ΟΗΕ, όχι της Ένωσης. Και βέβαια οι αυτοί που ασχολούνται με τα ανθρωπιστικά δεν τους άρεσε η στρατιωτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γι' αυτό και υπήρχαν οι πτώσεις επιφυλάξεις. Αυτό πάντοτε το, το δίλημα υπάρχει. Δηλαδή από τη μια θέλει κανείς να προστατεύσει με ενόπλου αυτού που δίνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Από την άλλη μεριά όμω, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτοί που δίνουν ανθρωπιστική βοήθεια εμπλέκονται πράκτο στην τοπική σύγκρουση και άρα επισύρουν τι επιθέσει των εμπολέμων. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αντιλαμβάνομαι ο κύριος Βανόρτεν Θέλει τον λόγο. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πού μπορεί να προσφέρει την αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα οποία εξετάσαμε αφορούν τα συμφέροντα κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της Αφρικής, δηλαδή του, του, που εκεί θα πρέπει να πρετανεύσει σταθερότητα. Και άκουσα τι είπε ο καθηγητή Κούπ όσον αφορά την ποικιλία, την, ε, το, πολυάριθμο των μεταβλητών ή των εμπλεκομένων. Οπότε δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο ευρωκεντρικοί στον προβληματισμό μα Και αν θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί, έχει, έχει ε, συνεργαστεί με την Αφρικανική Ένωση και κάνει εκπαίδευση και υποστηρίζει ε, αυτή την δύναμη επιφυλακής την Αφρικανική, τότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε. Πού έγκυται η προσθέμενη αξία από την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι να γίνει απαντήσει κανείς τώρα. Το αυτό το ερώτημα ως τροφή για σκέψη ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την κατάθεση πολύ δημιουργικών θα έλεγα θέσεων και βέβαια να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φιλοξενούμενους μας, τους εμπειρογνώμονες για την εξαιρετική παρουσίαση αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν που ήταν ολοκληρωμένες και πολύ συγκεκριμένες. Να υπενθυμίσω ότι αύριο συνεχίζουμε στις 9.30 στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με φιλοξενούμενον τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου. Σας ευχαριστώ.